Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Θα ομιλήσω ουγγρικά. Θα σας ζητούσα να φορέσετε τα ακουστικά σας, εκτός αν ομιλείτε ουγγρικά και καταλαβαίνετε τόσα λέω, ώστε να μπορούν οι διερμηνείς να διερμηνεύουν. Χάρη σας. Είναι διαθέσιμα τα πρακτικά της χρησινής συνεδρίασης. Υπάρχουν σχόλια σε σχέση με διαδικαστικά ίσως. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, τότε θεωρείτε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά της χρησινής συνεδρίασης. Σας